Okay, ladies and gentlemen, Καλά λοιπόν, κυρίε και κύριοι, ας αρχίσουμε την ε, συνεδρίαση της Επιτροπής. Ζητώ συγγνώμη και για την ελαφρά καθυστέρηση λόγω της κοινή ακρόασης δυο επιτροπών, των οποίων η μια είναι η δικιά μας. Μπορούμε να αρχίσουμε Σας υπενθυμίζω ότι είναι το πρώτο μέρος της συνεδρίας της Επιτροπής μας, δηλαδή και κλεισμένων των θυρών, που σημαίνει μόνο ευρωβουλευτές, γραμματεία και συνεργάτες των πολιτικών ομάδων. Ακόμα και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν επιτρέπεται να συμμετάσχει στη συζήτηση. Κλείνουμε δηλαδή τις πόρτες μας και για ένα